κάτι καλύτερα και μπορούμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε σε έναν οργανισμό που ήδη ασχολείται με τα σχετικά θέματα. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έχει κλείσει. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Περνάμε τώρα στην έκθεση Gross για τον ενιαίο χώρο μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος ομιλητής λοιπόν επαναλαμβάνει ο πρόεδρος είναι ο κύριος Γκρός. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στην Επιτροπή Μεταφορών συζητήσαμε ε, το, την Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές πολύ σοβαρά και υπήρξαν 413 τροπολογίες για να βελτιώσουμε τα θέματα που μας απασχολούσαν αλλά βρήκαμε μια καλή βάση καταλήγοντας σε 32 συμβιβαστικές τροπολογίες και είμαστε ε, ε, άλλωστε διαθέσιμοι προς συζήτηση και το υπήρξαν και οι συνάδελφοι γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες διότι όταν μιλάμε για μεταφορές μιλάμε για 10 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη μιλάμε για ένα μεγάλο ΑΕΠ μιλάμε για κάτι το οποίο ενδιαφέρει ε, τους πολίτες όλων των χωρών κάθε μέρα και γι' αυτό πρέπει να τεθούν τα ε, σωστά, ε, οι σωστές επισημάνσεις ή στη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια, για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, για το διοξίδιο του άνθρακος και ούτω καθεξής. Θέλαμε όμως να επισημάνουμε στο Συμβούλιο ότι πρέπει πιο γρήγορα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις για να καταργήσουμε τα σύνορα και στη συζήτηση αυτή υπήρξαν πολλές λέξεις μιλήσαμε για αποτελεσματικότητα αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να έχουμε σωστές συνθήκες εργασίας όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική πολιτική μεταφορών για την επόμενη δεκαετία γι' αυτό και διατυπώσαμε 31 σαφείς προτάσεις καταρχής για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών που έχουμε ε, χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο σε οδικά ατυχήματα πρέπει λοιπόν μέχρι το 2020 να μειώσουμε τουλάχιστον κατά 50% τα ατυχήματα αυτά επίσης ε, όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακος αποβλέπουμε με σε μία μείωση κατά 20% την επόμενη δεκαετία πράγμα το οποίο είναι δυνατόν με ένα μείγμα ενεργείας με μεγαλύτερη κινητικότητα με ε, μία ποικιλία μέσων μεταφοράς και ε, έτσι θα ζήσουν αύριο 80% των πολιτών με ε, διάφορα μέσα μεταφοράς πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο φιλικά προς τους πεζούς και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σκεφτόμαστε όμως και τον αέρα και το διοξίδιο του άνθρακος. Γιατί περιμένουμε το και καθυστερούμε τόσο πολύ όταν μπορούμε χωρίς επενδύσεις να έχουμε εξοικονόμηση κατά 20% διότι μιλάμε για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Θέλουμε να ανοίξουμε τις, μετα... τις ε, αγορές θέλουμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές μεταφορές, σκεφτόμαστε το οδικό σύστημα. Δεν θέλουμε η ε, μείωση των τιμών να οδηγήσει σε χειρότερες υπηρεσίες, θέλουμε να υπάρχει σωστή ανταμοιβή των υπηρεσιών για αυτούς οι οποίοι απασχολούνται στο χώρο. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό δίκτυο στην Ευρώπη για τις μεταφορές και να τονίσουμε θυμίσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να καταργηθούν διότι δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Αυτά είναι λίγα από τα παραδείγματα για το πώς διαβλέπουμε το μέλλον και κύριε Επίτροπε θα θέλαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσουμε στο μέλλον την διατύπωση του προγράμματος και να την εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δικός χάρτης για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών που έγινε δεκτός το 2011, καθορίζει το, το όραμά μας για μια αποτελεσματική μορφή ε, οργάνωσης του συστήματος μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ματιό Εγκρός όπως επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών για την προσπάθεια που έκαναν. Ξεκινήσαμε ήδη με την έκθεση του 2009 για την αηφορία στις μεταφορές. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη συμφωνία για τη σημασία που έχει να διατηρήσουμε ένα αποτελεσματικό τομέα στις μεταφορές. Οι μεταφορές στηρίζουν την οικονομία και την εσωτερική αγορά όλων των περιφερειών της Ευρώπης. Οι μεταφορές επίσης είναι ένας αποτελεσματικός οικονομικός χώρος, 10 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και άλλα 8 εκατομμύρια στην κατασκευή μεταφορικών μέσων. Είναι επίσης σημαντικά για την κοινωνική και την εταφική συνοχή. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένο ότι ο περιορισμό τη κινητικότητα δεν είναι σωστή εναλλακτική για να ε, εξασφαλίσουμε βιώσιμε μεταφορέ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπου για λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια και ε, καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών, προκειμένου να μην καταλήξουμε σε τόσο αρνητική εναλλακτική. Έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου κατά 60% μέχρι το 2050 σε σχέση με το 1990 και θεσπίσαμε και 10 στόχου που θα αποτελέσουν γνώμονα τη αξιολόγηση Προέδρου μέχρι το 2050. Φυσικά έχουμε και 40 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, τις τρέχουσες προκλήσεις και είμαστε προσιλωμένοι στο πρόγραμμά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2011 θα υλοποιήσει το 20% των πρωτοβουλειών της Λευκής Βίβλου και μάλιστα όχι τις λιγότερο σημαντικές. Θα συνεχίσω ε, ευχαριστώντας για την υποστήριξη της έκθεσής σας σε βασικές προτάσεις όπως είναι η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους μεταφοράς, η ενιαία ευρωπαϊκή εθέρες, η θαλάσσια γαλάζια ζώνη, ε, βιώσιμα σχέδια για κινητικότητες της πόλης και φυσικά η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς των μεταφορών. Όπως εξήγηλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας της, ε, θα υποβάλουμε πολύ φιλόδοξες προτάσεις το επόμενο, τον επόμενο χρόνο και για τους σιδηροδρόμους ε, θα, θα συμβάλλουμε στη δημόρφωση ενός ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου αλλά θέλουμε να συμβάλλουμε και στη δημιουργία πιο φιλοπεριβαλλοντικών οχημάτων και να θέσουμε προτεραιότητες για τεχνολογική καινοτομία προκειμένου να υλοποιήσουμε την πλήρη εσωτερήκευση όλου του εξωτερικού κόστους και να αποφύγουμε φορολογικές τρευλώσεις. Προσβλέπω σε συνεχή υποστήριξη και αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να δώσουμε σάρκα και οστά στις πρωτοβουλίες και προτάσεις της Λευκής Βίβλου. Ο κύριος Σόνικ έχει το λόγο. Φυσικά οι μεταφορές είναι ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ανάπτυξης και δημιουργεί πολλά εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης. Και φυσικά εξαρτώμαστε και από την διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό. Η διαχείριση των υποδομών και των μεταφορικών συστημάτων θα πρέπει να συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ελκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με την άρση των εμποδίων που ε, υπάρχουν στην απρόσκοπτη μεταφο... στις απρόσκοπτες μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό θέλουμε ε, έναν οδικό χάρτη για ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών και να μην ξεχνούμε τις τεχνολογίες που στηρίζονται σε μη ορυκτά καύσιμα και που ε, προκαλούν πολύ λιγότερα καυσαέρια η ανάγκη περιορισμού της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα και η προώθηση οικολογικών οχημάτων ή η εφαρμογή τεχνολογιών που ε, εξοικονομούν ενέργεια κατά την καύση είναι πολύ σημαντικέ προτάσει. Επίση, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία και τι νέε τεχνολογίε τη μεταφορέ. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ανάπτυξη των υποδομών στι νέε χώρε μέλη ε, και των οδικών μεταφορών μεταξύ άλλων κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα χρηματοδοτικά πλαίσια και προγράμματα εργασιών. Ευχαριστώ. Κύριος Κάρινς. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή ε, καλύπτει το 1 τρίτον της ε, κατανάλωσης ε, ενεργείας εις τις μεταφορές και εξ αυτού ουσιαστικά εξαρτάται από τις εισαγωγές. Γι' αυτό και οι μεταφορές εξαρτώνται υπερβολικά από τα, τις εισαγόμενες πρώτες ύλες. Οι εισαγωγές αυτές πρέπει να μειωθούν. Πώς θα το επιτύχουμε. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Καταρχήν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικά την ε, ενέργεια θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε βιοκαύσιμα και τέλος θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη πρόθεση της ηλεκτρικής κινητικότητας. Στηρίζω την έκθεση αυτή η οποία τονίζει την ε, εξάρτησή μας και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε στον τομέα των μεταφορών και σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής απουσία, ε, απουσιάζει, ευτυχώς γιατί δεν θα μπορούσα να προφέρω και το όνομά του. Ο μέθε επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Κοχ. Dieter Koch, ja. Ja. Herr Präsident, Herr Kommissar. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, για πολλούς ε, οι μεταφορές είναι ένα αναγκαίο κακό που ρηπαίνει ε, και θορυβεί στο περιβάλλον και η κατάσταση είναι μεν παράδεκτη αλλά είναι απαραίτητη για την λειτουργία της κοινωνίας μας, για την ευημερία μας και είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλους και ιδίως για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες που θέλουν να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς. Γι' αυτό και ε, χαιρετίζω τις διατάξεις και ρυθμίσεις της Λευκής Βίβλου για τα τρόπον ώστε να μην υπάρχουν αυθαίρετες ε, κινήσεις. Ο εισηγητής ε, κύριος Γκρός είναι έπαινος διότι μπόρεσε να διατυπώσει μία σωστή πολιτική και να καθορίσει στόχους χωρίς να αμφισβητήσει την τεχνολογία που διατίθεται. Ε, προσπαθεί να βελτιώσει τις προδιαγραφές για τη μεταφορά ατόμων, ε, ε, αγαθών, για το περιβάλλον, για τις συνθήκες εργασίας και για τις κοινωνικές ρυθμίσεις. Δεν τον βλέπω όμως να είναι αρκετά θαραλέως στην ρύθμιση ε, των ε, φορτηγών ε, αυτοκινήτων και βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει μία κατανομή των αρμοδιοτήτων διότι με το κείμενο αυτό μπορούμε να διατυπώσουμε στην Ευρώπη ελάχιστες προδιαγραφές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη κατά την διαδικασία διαδικασία της επικουρικής χορηγήσεως αδειών κατά τρόπον ώστε στο μέλλον να μην χρειαστεί να ξοδεύουμε πάλι πολλά χρήματα για να καταργούμε αυτά που εντωμεταξύ έχουν δημιουργηθεί. και τα φορτηγά αυτά θα πρέπει να σέβονται τα, τις επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Η κυρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρόταση, η Λευκή Βιβλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το 2050 είναι πολύ σημαντικό εγγραφό που δίνει κατευθύνσεις για την πολιτική μεταφορών. Είναι πολύ καλό υλικό και δημιουργεί και ένα πλαίσιο για τα βράχη μέσο και μακροπρόθεσμα βήματά μα. Απευθύνουμε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει συγκεκριμένου στόχου ε, για το 2020. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την τρέχουσα κατάσταση. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται σε προηγούμενα έγγραφα πολιτική και να ανταποκρίνεται, να αντικατοπτρίζει μάλλον την κατάσταση των υποδομών στα κράτη-μέλη. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει την ανάλυση τη μέχρι το 2013 το αργότερο. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχή και τα διάφορα μέσα και εργαλεία της θα πρέπει να εξασφαλίσουν εναρμόνιση των υποδομών των κρατών μελών με βάση τις αρχές της ασφάλειας και τη συμπερίληψη των εργασιακών συνθήκων των επαγγελματιών του κλάδου, γιατί ο κλάδος των μεταφορών απασχολεί περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ένα σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Το θέμα της ποιότητα της εργασίας, της κατάρτισης και της ασφάλειας στις μεταφορές είναι σημαντικά θέματα, γιατί οι μεταφορέ είναι τομέα που έχει άμεση συνέπεια στην καθημερινότητα και στην ζωή και ασφάλεια των πολιτών. Θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα λοιπόν και της ε, μακροπρόθεσμης πολιτικής και των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, στην ανάγκη πρόθεσης ε, βιώσιμων τρόπων μεταφοράς για όλες τις αποστάσεις και συμφωνώ ότι για τις μεγάλες αποστάσεις χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ελαστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας του και Πιστεύω ότι η πρόταση θα υποστηριχθεί από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, αγαπητέ Ματιό Γκρός. Αυτή ήταν εξαιρετική δουλειά που έκανες, διότι είπαμε υπήρχαν πέραν των 413 τροπολογιών και 30 τόσες συμβιβασικές τροπολογίες, πράγμα που δείχνει ότι όλοι δουλέψαμε σκληρά διατυπώθηκαν διάφορες ιδέες για διάφορα θέματα αλλά όλοι συμφωνήσαμε ότι οι μεταφορές είναι σημαντικές είναι η κινητήριος δύναμης ε, της ε, ενιαίας αγοράς χρειαζόμαστε ε, κινητικότητα για τους πολίτες και μπορούμε να πούμε ότι διεφάνει σαφώς όπως φαίνεται και στην έκθεση αυτή ότι χρειαζόμαστε όλα τα μεταφορικά μέσα. Θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη συχνότητα, αλλά για να μπορέσει να προωθηθεί ε, η ευρωπαϊκή αγορά χρειαζόμαστε όλα τα μεταφορικά μέτρα και αυτό τονίστηκε. Δεν υπάρχουν τόσα σημεία στα οποία διαφωνούμε. Ένα είναι τα μεγάλα φορτηγά. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές ομάδες αλλά είπαμε χρειαζόμαστε European Modular System δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο μήκος, μεγαλύτερο βάρος ορισμένοι δεν συμφωνούν αλλά λειτουργεί σε ορισμένα σημεία της Ευρώπης και τέλος για την, τους φιλελεύθερους θέλω να υπενθυμίσω μία τροπολογία την οποία προσθέσαμε την τελευταία στιγμή και θέλω να σας πω ότι το θέμα δεν είναι εδώ να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι σχετικά με τους σιδηροδρόμους αλλά να διαχωρίσουμε το δίκτερο από, τον, ε, ε, από την εκμετάλλευση και ε, ελπίζω ότι όλοι θα ακολουθήσετε την πρότασή μου. Σας ευχαριστώ και περιμένω με τα μεγάλου ενδιαφέροντος αύριο την, την ψηφοφορία. Ο κύριος Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον συνάδελφο Γκρός, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική συνεργασία και καταλήξαμε σε καλό αποτέλεσμα, διότι ε, χωρίς αλλαγή της κινητικότητας δεν θα μπορέσουν να υπάρξουν οι αλλαγές ε, στις κλιματολογικές συνθήκες και γιατί, διότι έχουμε επιτύχει μία μείωση κατά 34% στην ενέργεια και εντωμεταξύ στην, ε, ε, στις μεταφορές αυξήθηκαν οι εκπομπές κατά 13% πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι ε, γίνονται και καταστρέφονται αυτά τα οποία σε άλλους τομείς επιτυχάνονται με μεγάλες δαπάνες και μεγάλη προσπάθεια. Τώρα λοιπόν βρήκαμε μία συμβιβαστική λύση για να υπάρξει μία μείωση κατά 20% μέχρι το 2020 βάσει του 1990 και όχι του 2008. Το ξύναμε και θα παρακαλούσα όλα αυτά να υιοθετηθούν, να λειτουργήσουμε γρήγορα, να αντιμετωπίσουμε εσωτερικά όλους τους απάνες, να μην υπάρχουν υπεργολαβίες διότι η αεροπορικές αεροπορικές μεταφορές ε, επιδοτούνται από όλους τους πολίτες για την κεροζίνη. Έχουμε ε, υποχρεωτικές ρυθμίσεις για όλα τους σιδηροδρόμους και έχουμε και ε, δυνατότητες που έχουν εφαρμοστεί για τους αυτοκινητοδρόμους. Χρειαζόμαστε όμως και τα ποδήλατα και όλες τις δυνατότητες δεν δεν ε, πρέπει να μεταφέρουμε από το σιδηρόδρομο τις ε, μεταφορές στο δικό δίκτυο διότι όποιος δεν κατάλαβε το νόημα απατάτε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Μάτιου Γκρός για την εξαιρετική του δουλειά. Δυστυχώς όμως ε, εξακολουθεί να με ανησυχεί η βάση της έκθεσης, δηλαδή η λευκή βιβλία της Θέλω να είμαι δίκαιο ω προ την ε, Κομισιόν. Το έγγραφό τη κάνει μερικέ θετικέ ε, συστάσει ε, για τις ανάγκες ε, ε, σωστή διαχείρισης του συστήματος κλπ. Όμως η έκθεση αυτή έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Η Κομισιόν πιστεύει ότι η περισσότερη ρύθμιση και η περισσότερη παρέμβαση πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η απάντηση. Ε, αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη είναι ο βασικότερος παράγοντας των επιχειρήσεών μας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι τις πιέζουν και τις στενεύουμε ακόμα περισσότερο. Ε, η εναρμόνιση των κοινωνικών συνθήκων κλπ. θα ήταν παράλογες. Θα έπρεπε να καταργήσουμε τις ε, πειθαρχικές κυρώσεις και τις ποινικέ ε, και γενικότερα τις κυρώσεις. Η έκθεση επίσης καλεί σε μια αύξηση των διοδίων ε, στις οδικές μεταφορές. Αυτό δεν καταλαβαίνω πώς θα βοηθήσει την κινητικότητα. Το ίδιο ισχύει και με την απαγόρευση ε, της κυκλοφορίας στα κέντρα της πόλης αυτοκινητοχημάτων ε, με παραδοσιακούς κινητές εσωτερικής καύσης. Ε, ιδιαίτερα, είναι, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο στη σημερινή περίοδο οικονομικής ε, δυσχέρειας. Ε, η, γενικότερα η έκθεση ε, δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στι επιχειρήσει, υποστηρίζοντα την ανάπτυξη. Ε, ενώ αυτό το έγγραφο κάνει το ακριβώ αντίθετο, αποτελεί μια επιβάνηση επιχειρήσης. Ευχαριστώ. Ο κ. Τούσα. Η πολιτική τη απελευθέρωση και τη ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθιά αντιλαϊκή. Οι δημόσιε μεταφορέ ξεπουλήθηκαν στου μονοπωλιακού ομίλου μαζικέ απολύσει γενικευμένη εφαρμογή των ελαστικών μορφών απασχόληση και δραστικέ μειώσει των μισθών των εργαζομένων στον κλάδο εντατικοποίηση τη δουλειά των εργαζομένων και υποβάθμιση των κανόνων ασφάλεια με αποτέλεσμα την αύξηση των ατυχημάτων εκτείναξη στα ύψη των τιμών των εισιτηρίων και στα ανάβλα των εμπορευμάτων δραματική υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφοράς συγκοινωνιακό αποκλεισμό απομακρυσμένων υπηρετικών και νησιωτικών περιοχών οδυνηρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. η κατάργηση του καμποτάζ στην ελλάδα στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές ενώ συνοδεύτηκε με την προκλητική ενίσχυση των μεταφορικών ομίλων με πακτολό κρατικών επιδοτήσεων οδήγησε στον αποκλεισμό της απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές και τεράστιες αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων. με το ξεπούλημα του οσε ολόκληρες περιοχές πάβουν να εξυπηρετούνται σιδηροδρομικά και χιλιάδες εργαζόμενοι πετιούνται στον δρόμο. καθεστώς γαλέρας ισχύει και στις αερομεταφορές. το συμπέρασμα που βγαίνει για τους εργαζόμενους είναι ότι όσο κριτήριο θα αποτελεί η κερδοφορία των μονοπωλίων είναι αδύνατο να ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκέ ανάγκε. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκρός για την εξαιρετική του έκθεση. Ο τομέα των μεταφορών ε, εν γέννη είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι περιοχέ τη και του πολίτε τη Ευρώπη. Δημιουργεί θέσει απασχόληση και ενισχύει την ενιαία αγορά. Οι μεταφορέ μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στο στόχο τη Ευρώπη του 2020, ιδίω στου τομεί τη απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξης, έρευνας και περιβάλλοντος. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ορισμένα κράτη-μέλη υποτιμούν τη σημασία των μεταφορών και δεν ε, μεταφέρουν σε εθνικό δίκαιο οδηγίες και κανονισμούς εγκαίρως. Σε εποχές οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν προωθούμε επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να συνδέσουμε τις μεταφορικές υποδομές των παλαιότερων κρατών μελών θα πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές στην ανάπτυξη των υποδομών και η Ευρώπη χρειάζεται ένα ανταγωνιστικό σύστημα μεταφορών με βάση την αποδοτική χρήση των πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Στάσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φαίνεται πως τις ε, Βρυξέλλες, ένα, ο χάρτης για ένα ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών σημαίνει περισσότερα κονδύλια για τον τομέα των σιδηροδρομικών. Αλλά δεν είμαι κατά των σιδηροδρόμων, αλλά θα πρέπει να χορηγήσουμε περισσότερα κονδύλια σε αυτούς τους τρόπους μεταφοράς ε, από τις, τις οδικές και τις αεροπορικές. Δεν υπάρχει όμως κάποια αναλογία, δεν αναφέρονται οι υπόλοιποι τρόποι μεταφορών. Έχουμε τη στρατηγική του 2020, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν έχουν γίνει πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά τα δισεκατομμύρια επενδύσεων, τι αποτέλεσμα θα αποφέρουν. Νομίζω ότι η ελίτ των Βρυξελών θα ωφεληθεί, ενώ οι κοινοί πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν πέραν, ε, μάλλον παρά τις ε, σημαντικές ε, κρατικές επιδοτήσεις, το ποσοστό των συνδρομικών μεταφορών περιορίστηκε και βαίνει μειούμενο χρόνο με το χρόνο. Εδώ και δεκαετίες μιλάμε για στόχους σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Νομίζω ότι πρόσφατα ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των μεταφορών το παίρνουν οι οδικές μεταφορές και οι αεροπορικές μεταφορές. Αυτό δεν νομίζω ότι ωφελεί στο περιβάλλον. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική είναι απόλυτα εσφαλμένη. Χρειάζεται λοιπόν να διασφαλίσουμε την αντιστροφή της κατάστασης. Ευχαριστώ. Καταρχήν ο κύριος Κράμερ, για τον κύριο ε, ο κύριο Κράμερ έχει μια μπλε κάρτα για την κυρία Στάσεν. Δέχεστε κυρία Στάσεν. Πολύ ωραία. Κύριε Κράμερ, έχει το λόγο. Είπατε ότι δίνουμε προνόμιο στο σιδηρόδρομο. Ξέρετε ότι ο σιδηρόδρομος ε, πρέπει να πληρώνει όλη τη χρήση ηλεκτρισμού ε, ε, και βενζίνης, ενώ κάθε χρόνο στις αερομεταφορές υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν επιβαρύνσεις για κάθε μηχανή όθηση σιδηροδρόμου σε όλες τις σιδηροδρομικές γραμμές όταν υπάρχουν ε, διόδια στους αυτοκινητόδρομους συνήθως βαρύνουν ε, ε, περισσότερο τους οδηγούς επιβατικών οχημάτων και όχι τους οδηγούς των φορτηγών. Φαίνεται να είναι διπλάσια επιβάρυνση για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τους σιδηροδρόμους. Αυτό το έχετε λάβει υπόψη σας. Κυρία Στάσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κράμερ, εμείς έχουμε διστάμενες απόψεις, αλλά οι σιδηρόδρομοι συνεχίζουν να επιδοτούνται και οι υποδομές, οι οδικές, αλλά και οι αεροπορικές είναι αυτές που πληρώνουν το τίμημα. Ευχαριστώ κύριο Σπέρκαλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε ε, ε, διάφορους κανόνες ε, για τις ροές μεταφορών σιδηροδρόμου για τομείς που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ματιό ό ως εισηγητή, υπέβαλε εξαιρετικέ προτάσεις και μιλάει για τις ε, συνδυασμένες μεταφορές ε, και τις συντροπικές μεταφορές Μιλάμε για μέσα μεταφορών για όλες τις χώρες και για όλες τις περιφέρειες και δεν ε, μπορούμε ακριβώς τα ίδια μέτρα να μεταφέρουμε σε όλες τις ε, περιοχές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τα γίγκα ε, οχήματα για, τις, για μεγάλους όγκους μεταφορών μπορούν να αντικαταστήσουν φορτηγά. Κατά τη γνώμη μου για τη χώρα μου, την Αυστρία, θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ελάφρυνση των επιβαρύνσεων με τέτοιου είδους μέτρα, με υποδομές που πρέπει να είναι σωστά προσαρμοσμένες με ε, τις οδούς διαμετακόμισης για τις οποίες χρειάζεται να διατεθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Με την ε, τροπολογία που έχω κάνει στο σημείο 26 προτείνω να μην υπάρχει ε, ευρωπαϊκή έγκριση για τα ε, γίγα ε, φορτηγά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν σε κάθε κράτος μέλος αν θα δίδουν έγκριση για αυτά τα μεγάλα, ε, μεγάλου όγκου οχήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μεταφορές βιώσιμες και υφόρες για τον χώρο των Άλπαιων και για την Αυστρία θα μπορούν τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ελεύθερα εάν αυτά τα μέσα μεταφορών θέλουν να τα επιτρέπουν στο δικό τους δίκτυο ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαλκαντράουι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η, οχι ευχαριστω ευχαριστω κυριε σαλκαντραουι κυριε προεδρε κυριε επιτροπε κυριες και κυριοι η σημαντικη αυτή είναι πολύ σημαντική για το Κοινοβούλιο διότι δίνει την κατεύθυνση των εργασιών μας για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Έχει κατορθώσει να πετύχει και σωστούς και κατάλληλους ε, ε κατάλληλες προτάσεις ε, και συνεργασίες ε, κατά τα επόμενα χρόνια νομίζω δεν μπορούμε να απελευθερώσουμε το τομέα των μεταφορών και ταυτόχρονα να μην πράξουμε τίποτα προκειμένου να λάβουμε υπόψη όλες τις κοινωνικές πτυχές του ζητήματος. Ως εκ τούτου λοιπόν το 2013 η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια σε ανάλυση των ε, κοινωνικών συνθήκων σε όλους τους ε, μεταφορικούς κλάδους και αυτό προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συνθήκων εργασίας για όλους τους εργαζομένους και να καταστήσουμε και ελκυστικό τον κλάδο. Εξάλλου χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας πως θα υπάρξει και ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την οικονομία και για το περιβάλλον εάν δεν εξευρεθούν λύσεις αποτελεσματικές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα πολιτικής όπως και ένα μείγμα ενεργειακό, εναλλακτικές τιμές για τις ε, νέες τεχνολογίες, ε, για νέα καύσιμα κλπ. Ευχαριστώ πάνω στον εισηγητή. Τώρα σε ό,τι την ε, διατροπικότητα ιδιαίτερα στον τομέα των σιδηροδρόμων αλλά και στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών διότι ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να οδηγήσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης βλέπουμε ότι το θαλής ε, έχει ανάγκη από διαφορετική σήμανση για λόγους ασφαλείας πόσο ε, χρειάζεται να διασχίσει τρεις διαφορετικές χώρες. Άρα λοιπόν πολλά θα πρέπει να γίνουν και για την εναρμόνιση στον τομέα της σήμανσης. Πάντως η έκθεση αυτή αποτελεί ένα καλό σημείο αφιτερίας για την προσεχή χρονιά. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Γκρόσου για την εργασία του δεν ήταν διόλου εύκολο να βρεθούν οι κατάλληλες ισορροπίες. Περίπου 400 τροπολογίες ε, κατατέθησαν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία και να πετύχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο δαπανών παράλληλα με την του περιβάλλοντος η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά αποθετικά στοιχεία. Τονίζει ότι η ανάπτυξη των υποδομών στα κράτη-μέλη είναι κάτι το απαραίτητο. Μιλάει επίσης και για την ενιαία, ενιαία αγορά στον τομέα των μεταφορών. Πάντως η ομάδα μου βρίσκει δύσκολο να μπορέσει να στηρίξει όλες τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν στο κράτη μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ακόμα φορά επικαλούμαστε θεμητούς στόχους, αλλά επιδιώκουμε κάτι διαφορετικό. Η έκταση αναφέρεται σε στόχους περιβαλλοντικούς, ενέργειακή αποδοτικότητας, μείωση κατανάλωσης του άνθρακα, διαλειτουργικότητας, όλα καλά. Αλλά τελικά φαίνεται, διαφαίνεται τι πραγματικά επιδιώκει. Για μία ακόμα φορά επιμένουμε στην απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση, ο, οτιδήποτε μπορεί να δώσει κέρδος, με βλάβη βέβαια για τους ε, χρήστες, για τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους και για τις ε, εθνικές οικονομίες που απο, χάνουν ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξή τους. Κάθε κράτος έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες εξαιτία των ιδιαιτεροτήτων του και της σχετικής του ανάπτυξης. Το ερώτημα είναι ε, ποια συμφέροντα θα εξυπηρετήσει αυτή η ενιαία πολιτική μεταφορών τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών πολιεθνικών ε, που θέλουν ε, να πνίξουν τις αγορές με τα προϊόντα τους ε, γρήγορα και με χαμηλό κόστο και σίγουρα αυτά τα συμφέροντα είναι διαφορετικά από τα συμφέροντα των λαών που όπως, συμβαίνει στην Πορτογαλία με το πρόγραμμα του Διεθνούς Ταμείου αντιμετωπίζουν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Κάντσιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αύριο θα υιοθετήσουμε αυτή τη στρατηγική για το μέλλον των μεταφορών αλλά έχουμε ήδη τάπητος κάποιες νομοθετικές πράξεις συγχαρητήρια στον εισηγητή που μέσα σε τρεις μήνες κατόρθωσε να συντάξει ένα έγγραφο το οποίο μας κρατά δεμένους για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Η δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς στον τομέα των μεταφορών. Τα τεχνικά εμπόδια ε, αποθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και δεν καταλήγουν σε μείωση των κόστους ε, και του τμήματος το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές. Μετά από 25 χρόνια από την ψήφιση της ενίας πράξης υπάρχουν φραγμοί για, που παρεμποδίζουν αυτόν τον κλάδο να αναπτυχθεί. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας διότι αυτή η νέα αγορά είναι ένα μέτρο για την ε, ανάπτυξη της οικονομίας. Σκέφτομαι το άνοιγμα των αγορών, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημιουργικής αγοράς και την εφαρμογή της τεχνολογίας RTM σε όλο το δίκτυο. Οι υποδομές αναφέρθηκαν, αυτές οι ε, διασυνοριακές ε, κατά προτεραιότητα και η σύνδεση ανάμεσα στους, στα διάφορα δίκτυα. Οι υποδομές ε, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με τα κονδύλια τα οποία έχουμε προβλέψει. Τα PPP και οι εκπομπές, ε, και η έκδοση ε, ομολόγων σχεδίων νομίζω ότι είναι ουσιαστικά αυτά τα οποία ονομάζουμε project bond θα πρέπει να μας επιτρέψουν να πάμε παραπέρα, να λάβουμε υπόψη όλα τα θέματα της ε, οδικής ασφάλειας ε, και την διάδραση μεταξύ τους ε, εθέρες και ο πυλώνας Σέζαρ θα πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει ταυτόχρονα όμως να υπάρχει μια ε, ενιαία διακυβέρνηση. Ακούσαμε από τον Επίτροπο ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρξουν φιλόδοξε προτάσεις. Πράγματι εμεί ε, προσβλέπουμε σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Ulfskog. κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε. Η έκθεση ασχολείται με μια σημαντική ανάγκη του τομέα των μεταφορών. Γιατί δεν κάνουμε κάτι για να συνδυάσουμε μακροπρόθεσμες μακρόπνοες επενδύσεις και ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε την μακρόχρονη ανεργία. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών θα πρέπει να ε, προωθηθούν έτσι ώστε να μειωθεί να μειωθούν εκπομπές διοξείδου του άνθρακα και ταυτόχρονα γίνουν πιο φτηνές οι μεταφορές. Εξακολουθούμε να έχουμε στόχο για την ε, μείωση ε, του διοξιδίου του άνθρακα 20% μέχρι το 2020 ε, και θα πρέπει να να πάμε και ακόμα πιο μακριά. Ας δούμε τι, τι σημαίνει σε αυτό το τομέα. πρέπει να δούμε τον ανταγωνισμό και το κοινωνικό dumping διότι αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους τομέα και ταυτόχρονα οδηγεί σε ατυχήματα και χαμηλές, και μειώνει τα στάνταρ της ε, ποιότητας. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις λοιπόν, χρειάζεται να βελτιώσουμε την ασφάλεια και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να βλέπουν τη διαφορά όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και οι χρήστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βλάσακ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κατάργηση των φραγμών ε, στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών ε, εμπορευμάτων και ατόμων είναι προτεραιότητα για μας. Γι' αυτό και είναι απαραίτητος αυτός ο ενιαίος χώρος και χρειαζόμαστε άξονες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα πολυτροπικό δίκτυο. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σωστό το ότι η Λευκή Βίβλος αναφέρει πολλές φορές τις διαφορές που υπάρχουν στις υποδομές ε, σε χώρες της Ανατολικής και της Δυτικής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένα μέτρα μέσα στη Λευκή Βίβλο για να αντιμετωπιστούν ακριβώς αυτές οι διαφορές. Νομίζω ότι η Επιτροπή δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα της πολιτικής στον τομέα αυτό. Περίμενα συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων, τα οποία θα έπρεπε ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως και πάλι τα ίδια κράτη-μέλη θα έχουν τις υψηλότερες επιδοτήσεις ε, ε, και ενισχύσεις παρότι οι χώρες αυτές λαμβάνουν 10 ε, δισεκατομμύρια που θα έπρεπε να πάνε προς πιο φτωχές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και τόσο ευρύ θέμα όπως η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές θα είναι πολύ δύσκολο να τα συνοψίσουμε ε, σε ένα σύντομο κείμενο. Βλέποντας ε, το κείμενο στο οποίο κατέληξε ο εισηγητής μας, δεν μπορούμε παρά να τον συγχαρούμε, γιατί από πολλές εκατοντάδες τροπολογίες κατόρθωσε να καταλήξει σε ένα πολύ καλό, συνεκτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι θετικό για τις μεταφορές του μέλλοντος, για την ασφάλεια, για την ενέργεια και για την τεχνολογία. Χαιρετίζω τα βασικά ζητήματα που αναφέρει σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, με τα κοινωνικά πρότυπα ε, και αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένων των ελλείψεων στον τομέα των μεταφορών, κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να αποφύγουμε μελλοντικέ συμφορήσεις των μεταφορών ε, στο μέλλον. Περαιτέρω άνοιγμα για το καμποτάζ και για τις οδικές μεταφορές υπό την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι πολύ σημαντικό να γίνουν Επίσης ε, χαιρετίζω το ότι αποδίδεται μεγάλη προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια. Η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο είναι ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει σοβαρά και στο μέλλον. Στις διατροπικές μεταφορές θα μπορούσαμε να ε, πούμε πολλά πράγματα και θεωρώ τη συζήτηση για τα Giga Liner ε, ως μια συζήτηση που δεν είναι η καλύτερη ε, λύση. Υπάρχουν θέματα και τεχνικής εναρμόνισης και ανταγωνισμού που πρέπει να επιληθούν και με την έκθεση αυτή ελπίζω ότι εκφράζονται οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου και θέλουμε να επιτύχουμε μέχρι το 2020 τους στόχους μας για να γίνουν οι προτάσεις μας πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παχνιό. Κύριε εισηγητά κύριε Επιτροπέ. Καταρχήν συγχαρητήρια στον εισηγητή για την συνένεση που εξασφάλισε. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την κυρία Σενάλοβα, η οποία οποία αποφάσισε να μην ζητήσει την ε, απελευθέρωση των υπηρεσιών λιμένος σε αυτό το κείμενο. Ε, θέλω να σας πω το εξής το λεπτό που μου μένει. Ε, από την υιοθέτηση του 2000, το 2001 του Λευκής Βουλίου για τις Μεταφορές έγιναν πολλές αλλαγές. Παρόλες τις προσπάθειες διαπιστώνουμε ότι 10 χρόνια μετά οι μεταφορές εξακολουθούν να μην είναι βιώσιμες. Οπότε πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής 28 Μαρτίου του 2011 ε, δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη. Και με μετά τον οδικό χάρτη που θα υιοθετήσουμε αύριο, ελπίζω στο μέλλον να υποβάλλετε πιο συγκεκριμένε προτάσει, για παράδειγμα επί της μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% σε οδικές μεταφορές, για την εφαρμογή τη αρχής ορυπαίνων πληρών σε όλες τις μεταφορές κλπ. Είπατε πρόσφατα ότι μέχρι το 2050 πρέπει τα κράτη-μέλη να ε, κινητοποιήσουν 1,5 ε, 1500 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ε, πώς θα επίσης θα ανταποκριθούμε στον οδικό χάρτη και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση την οποία ζητάτε στα κράτη-μέλη. Additional... Κύριε Φώστερ, έχετε ένα ακόμα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ένα ε, βιώσιμο τομέα μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρώπη. Αλλά χρειαζόμαστε την κατάλληλη πολιτική μεταφορά για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητά του, ε, απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ασφαλώς ένα μακρόπνο όραμα για την πολιτική μεταφορά και να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη του τομέα θα είναι βιώσιμη. Και πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να συνδράμουμε τον κλάδο για να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Όμως με ανησυχεί το ότι η έκθεση δεν είναι ισόρροπη. Ε, σαν να προσφέρει μόνο μία λύση για τη βελτίωση της ε, βιωσιμότητας των μέτρων μεταφορών. Δηλαδή νομοθεσία, νομοθεσία και ακόμα περισσότερη νομοθεσία. Ε, είναι υπερβολικά στενή αυτή η λύση και υπερβολικά παχθής θα οδηγήσει σε υπερβολικέ δαπάνε σε εθνικό και κοινωτικό επίπεδο. Από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα, γιατί να μην δούμε και άλλε αναλυτικέ λύσει. Για παράδειγμα, την, ε, ε, τις, ε, το να μοιραστούμε τι κοινέ πρακτικέ. Πρέπει να μάθουμε από άλλου ε, κλάδου για την μείωση του ίχνου διοξιδίου του άνθρακα. Για παράδειγμα, το μέσο των αέριων μεταφορών έχουν έχει κάνει σημαντικέ προσπάθειε για τη βελτίωση τεχνολογία. Ε, αλλά αυτό δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου. Και βέβαια έχουμε και τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό ε, που, θα, ε, που υποστηρίζει πάρα πολύ η ομάδα μου θα ήταν ε, μια, μια λύση για να αντιμετωπίσουμε την κυκλοφορία στους εθέρες. Τέλος, να πω ότι αν θέλουμε να είμαστε λογικοί θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες ε, που θα μειώσουν το άχθος ε, στον κοινοτικό προπολογισμό, θα ενθαρρύνουν τον κλάδο και κυρίως θα βοηθήσουν τους ε, εκλογείς να μετακινούνται πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόζα. Ε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Νομίζω πως ο κύριος Γκρός έκανε εξαιρετική εργασία και είμαι της άποψης ότι ε, έφτασε με την κατάλληλη απάντηση σχετικά με το μέλλον των ε, μεταφορών. Επανειλημμένα στις ε, δηλώσεις μου είπα ότι χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο φιλικό στο περιβάλλον και αποτελεσματικό μεταφορικό σύστημα. Ένα όμως θεμελιώδες ζήτημα είναι πως ε, θα πρέπει να έχουμε και μια χάρτα για τα δικαιώματα των ε, επιβατών για κάθε τρόπο μεταφοράς, ε, για κάθε μέσο μεταφοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή διότι τόνισε το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία διότι Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη είναι, είναι μια <clears throat> ήπειρος ε, και αποτελεί από κοινωνίες που γυράσκουν και καταλαβαίνετε ότι θα αντιμετωπίσουμε όλο και περισσότερο τα θέματα των ΑΜΕΑ στις μεταφορές. Στο προσεχές μέλλον θα δούμε οι ανάγκες αυτών των ατόμων να πολλαπλασιάζονται κατά την χρήση των μέσων μεταφορών. Είμαι της γνώμης λοιπόν πως ε, στον έκθεση περιλαμβάνεται ένα σαφές μήνυμα να τονίσω για μια ακόμα φορά πως θα πρέπει να διασφαλίσουμε το 2012 η Κομισιόν να λάβει υπόψη της όλα αυτά τα στοιχεία και να τα συμπεριλάβει σε μια πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος αγορτή, ο κύριος Ερτούγκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τις Μεταφορές όπου υποβάλλονται προτάσεις για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και στόχοι για τα επόμενα 20, 30 και 40 χρόνια είναι ένα πολύ μακροπρόθεσμο σχέδιο. Θέλει πολύ μακροπρόθεσμους στόχους. Οι μεταφορές χρειάζονται μακροπρόθεσμους στόχους. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή. Βλέπουμε τους φιλόδοξους στόχους της Επιτροπής, τους οποίους ε, επικροτώ, και βλέπουμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, με καλύτερες τεχνολογίες, βελτίωση των μεταφορών μέσω της διατροπικότητας, εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και κυρίως οι μεταφορές θα πρέπει να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι πολύ θετικά όλα αυτά τα οποία ε, έχει κατά νου η Επιτροπή. Βλέποντας τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου Και όσον αφορά τις εσωτερικές οδούς ε, ναυσιπλοείας, θα πρέπει να προωθήσουμε την ναυσιπλοεία σε ποταμούς όπως ο Δούναβης και συμφωνώ ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, να προσαρμοστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο με τις ανάγκες των ε, πλωτών μεταφορών. ο εισηγητής ήταν πρόθυμος να λάβει υπόψη του πολλές τροπολογίες και ένα σημείο ακόμη το θέμα των 300 χιλιόμετρων πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε περάσει πάντως και έτσι όπως είναι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ευχαριστώ πολύ Τώρα περάσαμε στο γύρο του Catch the Eye υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τον λόγο θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι θα σας διακόπτουμε μόλις φτάσετε στο λεπτό. Κύριο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξωτερική δουλειά του υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα την ετήσια αξιολόγηση που θα επιτρέπει να παρακολουθούμε τις, την πρόοδο και αν είναι δυνατόν και αν χρειάζεται να προσαρμόζουμε τους στόχους στην πραγματικότητα των κρατών μελών έτσι ώστε ε, να επιτευχθούν οι στόχοι αυτή τη φορά. Να επιγραμμίσω επίσης ότι χρειάζεται να συντονίσουμε τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων με το Ταμείο Συνοχής και να καταστήσουμε σαφές ποια είναι τα σχέδια που ε, μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Σε ό,τι αφορά τις από ε, απόκεντρες περιοχές, για πρώτη φορά δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτές. Αντίθετα με τη Λευκή Βιβλίο του 2001. Η εσωτερική αγορά όμως εκτείνεται και σε αυτές τις ε, περιοχές. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ο λόγος στην κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεσή του για τον τομέα των μεταφορών. Θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις για το άνοιγμα της αγοράς δεν θα οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ ούτε σε ιδιωτικά μονοπόλια που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε επιδείνωση των κοινωνικών συνθήκων και των συνθήκων εργασίας καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Τα νέα κράτη-μέλη έχουν ανάγκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και στα επόμενα ε, πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια. Μέχρι το 2020 το δίκτυο μεταφορών στα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, γεφυρωθεί και να κλειστούν τα κενά που υπάρχουν τώρα στις μεταφορές μεταξύ ανατολικών και ε, δυτικών χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακόπτεται το μικρόφωνο. κύριε Σάσκον η Λευκή Βήλωση του 2001 χαρακτηρίζεται από την απουσία πολιτικής βούλης των κρατών μελών. Γι' αυτό το ε, λόγο η πρόκληση είναι η εναρμόνιση και η απλοποίηση της κοινωνικής νομοθεσίας, στην ασφάλεια, στις εργασιακές συνθήκες, στο χρόνο οδήγησης, εσωτερικοποίηση του κόστους και βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες. Μέσω της ενίσχυσης των, των θαλάσσιων οδών, ε, της ε, ε της, ε, πολυ, ε, των πολυτροπικών μεταφορών και λοιπά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος με λιγότερους θανάτους, περισσότερη καινοτομία και πιο ε, ενοποιητική. Αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη αποφασιστικότητα από τα κράτη-μέλη. Δέκα χρόνια μετά τη Λευκή Βίβλο χρειαζόμαστε επίγοντα μέτρα, διότι διαχειριζόμαστε μια κρίση της μεταφορά των μεταφορών στην Ευρώπη. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Ιζεμπέλ Γιού. Εκτός μικροφώνου. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί φίλοι, η διάσκεψη του Ντέρμαν μόλις έκλεισε, γλιτώσαμε την πνιγμό, αλλά ε, το, πετύχαμε κάποια αποτελέσματα. Αυτή η λευκή δήλωση για μας, κύριε Πίτροπε, είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να μπορούμε να κάνουμε κάτι στην ε, τομέα του μεταφορών. Διότι νομίζω ότι η ενεργειακή απόδοση, ο τρόπο ε, το να δημιουργήσουμε καινοτομίε, ανάπτυξη άλλων μέσων, τρόπων μεταφορά, η ενεργειακή απόδοση. Το είπα ότι ήδη απέδωσε. Έχουμε δημιουργήσει θέσεις εργασίας, ε, νέους τομείς, ε, νέους κλάδους. Σας καλώ λοιπόν κύριε Επίτροπε να είσαστε ιδιαίτερα φιλόδοξος και ε, θαραλέος. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν μέσω από, με, αυτήν την λευκή βίβλο να κάνετε περισσότερα και αποτελεσματικό στον τομέα των μεταφορών, να αναπτύξετε τις καινοτομίες, νέους κλάδους, πιο καινοτόμους αλλά και νέες πρακτικές, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας και αυτό θα, είναι αποτέλεσμα, θα, είναι, θα έχει ως αποτέλεσμα το καλύτερη διαβίωση των πολιτών. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος σας, ε, Ιζαμπέλ, ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών είναι μια πολύ σημαντική φιλοδοξία και γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις εθνικέ διατάξεις κατά τον αντίστοιχο τρόπο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο με την απαραίτητη εναρμόνιση χωρίς βέβαια να υπάρχουν περιττοί περιορισμοί. Οι κοινοί ε, κανόνες θα πρέπει να προωθήσουν τον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών είναι και η πηγή του ενός τετάρτου των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε στην πολιτική μας υπέρ του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέλτσερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τωρινή Λευκή Βίβλο υπάρχουν οι στόχοι για τα επόμενα δέκα χρόνια και τα επόμενα χρόνια για να έχουμε αποτελεσματικά προγράμματα από τις Βρυξέλλες Υπάρχει ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όλα αυτά τα οποία πολύ συχνά αποτελούν πολύ περιορισμένες πρόοδους. Υπάρχουν στη Λευκή Βίβλο και πολύ φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα, για τη δημιουργία ενός ε, χώρου χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Ε, θέλουμε αηφόρο τομέα μεταφορών για να μπορούμε να έχουμε και βιώσιμη οικονομία και όλα αυτά συνδέονται βέβαια και με το κλίμα και με τις ανάγκες των πολιτών για κινητικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μέλτσα. Ο κύριος Μίκολας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μεταφορών και η συνάρτησή της με την καθημερινή ζωή των πολιτών και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικά θέματα για όλους μας. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό εργαζομένων, για 10 εκατομμύρια απασχολουμένους. Ε, είναι ένας τομέας που προωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε ποιότητα υποδομών και ενίσχυση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται καλή διατροπικότητα και διαλειτουργικότητα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ κρατών μελών, δεν θα πρέπει στα σύνορα να παρακολύονται οι μεταφορές και δεν θα πρέπει να είναι σε ανταγωνιστική θέση τα μέσα μεταφορών, θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τις περισσότερες από τις ε, προτάσεις της ε, Λευκής βιβλού, λέει ο κ. Μπαλιώτης γιατί έχουν ως ε, στόχο ε, τη, τη βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών. Το σημαντικό είναι να συνδεθούν όλα τα μέσα μεταφοράς στα κράτη-μέλη, όλοι οι τρόποι μεταφοράς στα κράτη-μέλη και γι' αυτό χρειάζεται να αναπτύξουμε το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών. Χρειαζόμαστε να απορροφήσουμε καλύτερα ασφαλώς τους κοινωτικούς πόρους, τα κοινωτικά κονδύλια. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Ε, άλλο ζήτημα είναι να συνδέσουμε ε, τα δικά μας στήματα μεταφορών με αυτά τρίτων χωρών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τα σημεία μετάβασης ε, στα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με τους, κυρίου, με τους πιο σημαντικούς γειτονές μας. Ευχαριστώ κύριος Λούχαν. Κύριε Πρόεδρε, οι μεταφορές δεν περιορίζονται σε μία χώρα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ισχυρή διεθνή συνεργασία ώστε οι δράσεις μας να είναι αποτελεσματικές σε αυτόν τον τομέα. Δυστυχώς ένα από τα βασικά ε, εμπόδια για τη δημιουργία μιας ενιαίας ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών είναι οι σημαντικές ε, διαφορές ε, στις υποδομές ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι οι περιφέρειες που υστερούν θα πρέπει να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται αρκετά ώστε να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Η βελτίωση των υποδομών και της πρόσβασης ε, θα συνεισφέρει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών των περιοχών και προφανώ έμεσα στην ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούχαν και ευχαριστώ όλου όσοι προσπάθησαν να παραμείνουν εντό του χρονικού πλαισίου. Να δώσω το λόγο τώρα, αφού ολοκληρώθηκε το Catch the Eye, να δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Επίτροπο κ. Κάλλας, προκειμένου να σχολιάσει τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Κύριε Κάλλας, για το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι κατανοητά όλα αυτά και από όλε τι ε, παρατηρήσει καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι ο τομέα των μεταφορών και πόσε πολλέ είναι οι λεπτομέρειε που πρέπει να βελτιωθούν σε αυτό τον τομέα. Ακούσαμε και πολλές διστάμενες απόψεις για τον τομέα των μεταφορών. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι ε, λίγες οι ρυθμίσεις και πρέπει να τις βελτιώσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Χρειαζόμαστε αυτόν τον ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο μεταφορών. Αν τα έργα δεν προχωρούν όσο γρήγορα επιθυμούμε, πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Εγώ πιστεύω πως σίγουρα και δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι και να προσπαθούμε να ολοκληρώνουμε το έργο μας. Δεν έχω πολύ χρόνο για να αναπτύξω όλες τις θέσεις μας επ' αυτού. Πάντως έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ήδη έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις και σε σχέση με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Κάνατε μια συζήτηση για την αναδιατύπωση του πρώτου πακέτου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και είδατε πόσα πολλά θέματα υπάρχουν σε αυτό τον κατακαιρματισμό, κατακαιρματισμένο τομέα των μεταφορών, πόσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και πόσα διαφορετικά συμφέροντα. Πολλοί από εσά αναφέρατε ότι αυτή η λευκή βίβλος ε, έχει την πρόθεση να αυξήσει το επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων. η βιομηχανία παραγωγής σιδηροδρομικού υλικού και υλικού των μεταφορών διαμαρτύρεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές διατυπώσεις και διαδικασίες στα κράτη-μέλη που είναι χρονοβόρες ε, και δαπανηρές. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης, ε, πράγμα το οποίο δεν θα σημαίνει περισσότερα, αλλά λιγότερη, ε, λιγότερες ρυθμίσεις. Θέλουμε να μειώσουμε τις διατυπώσεις για τα σκάφη. Περιορισμός λοιπόν και πάλι των ρυθμιστικών διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφορών όσο το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικό. Το θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, καθώς και το θέμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, καθώς και την εξάρτηση από τα ε, ρηκτά καύσιμα. Ε, θέλουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα για να μην απογοητεύσουμε τον κλάδο, τους πολίτες, τα κρατη όλους τους ενδιαφερομένους. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη πρόταση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και η διευκόλυνση Connecting Europe που είναι διαφορετική σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις για τους σιδηροδρόμους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πώς να υπερβούμε ε, τον εθνικό κατακαιρματισμό αυτών των τρόπων μεταφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε τη συζήτηση δίνοντας τον λόγο στον εισηγητή τον κύριο Γκρός. Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και προς συνάδελφο συναδέλφους θα ήθελα να πω ότι ε, ε, οι μεταφορές είναι ένας τομέας στους οποίους λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και για τους αναπήρους και για τις οικογένειες και για τους ηλικιωμένους ε, δεν ε, κάνουμε νομοθεσία χάρη της νομοθεσίας και οδηγίες χάρη των οδηγιών. Θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνο όταν ε, είναι απλούστερες οι ευρωπαϊκές διατάξεις από τις 27 διατάξεις των κρατών μελών. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργη η στάση των συναδέλφων που λένε ότι η Ευρώπη μας δυσκολεύει τη ζωή. Μα, ο σκοπός μας δεν είναι να δυσκολεύσουμε τη ζωή των πολιτών, αλλά διευκολύνουμε με μια κοινή διάταξη αντί των 27. πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση και ήδη το ακούσαμε ότι πολλοί πιστεύουν ότι ένα προϊόν βελτιώνει το μέλλον ε, και αυτά τα γιγαντιαία φορτηγά, τα gigalines, για άλλους είναι πανάκια και για άλλους καταστρέφουν ε, τα πάντα. Σε πολλές ε, χώρες τα θεωρούν απαραίτητα, στην Αυστρία τα θεωρούν απαράδεκτα. Δεν θα μπορούσαμε με τέτοια αντιμετώπιση λοιπόν να καταλήξουμε σε κοινέ οδηγίες Κύριε Επίτροπε, θα ξεκινήσουμε αύριο την δουλειά ε, ε, ε, στην πράξη και κάθε μέρα και κάθε χρόνο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τις μεταφορές γιατί για μας είναι σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα μέσα για την οργάνωση των μεταφορών και αναχώρα και αναπεριφέρεια και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μαζί με την Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι όλες οι προσπάθειες και στα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορούν να βρουν μια λύση με την διαλειτουργικότητα και τη διατροπικότητα και τις συνδυασμένες μεταφορές και ε, αυτό το οποίο λέμε εδώ δεν είναι απλώς θεωρητικά αλλά από αύριο θα τεθούν σε λειτουργία και στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Η, ψηφο... η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30 το πρωί.